Il Presidente. Buongiorno colleghe e colleghi. Καλημέρα συνάδελφοι. Στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε την ε, ε, έκθεση Κιν Κακάλ ε, σχετικά με την ε, ουσιαστική εφαρμογή των θεμελιών δικαιωμάτων μετά την άρχιση ισχύ ε, της Συνθήκης Λισαβόνας. Το λόγο έχει η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας ε, έχει σε συνέπεια κοινοτικές αρμοδιότητες νέες κοινωτικές αρμοδιότητες, μια, ένα όραμα για μια ε, δυνατή Ευρώπη ε, και αυτό αφορά και την προστασία των θελειωδών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν, αντίθετα από ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, η αιτήσια έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, σχετίζεται με αυτή τη νέα νομική βάση για τις ενισχυμένες εξουσίες και αρμοδιότητες και εξετάζει τη νέα κατάσταση. Ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να υιοθετηθεί νέα προσέγγιση, μια σφαιρική προσέγγιση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από τον Δεκέμβριο του 2009 η προστασία των ε, ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων βασίζεται σε διάφορους πυλώνες. Πρόκειται για το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που γίνεται δεσμευτικός με την έγκριση της Συνθήκης Λισαβόνας που είναι σήμερα ένα σημείο αναφοράς για την κοινοτική νομοθεσία. Ένας άλλος βασικός πυλώνας είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ε, όπου είναι μέλος ε, συμβαλόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει μέλος. Ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, βεβαίως ε, κατοχυρώνονται και από τα συντάγματα των κρατών μελών. Αυτό είναι άλλος ένας βασικός πυλώνας. Υπάρχει νέο χαρτοφυλάκιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ομάδα εργασία στο Συμβούλιο και οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στην ε, αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία ε, των ε, υπαρχών των μηχανισμών και οργάνων. Είτε πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων, είτε για την υιοθέτηση εφαρμοστική νομοθεσία, είτε για την συλλογή ε, δεδομένων. Ε, δεν θα πρέπει όλα αυτά τα όργανα και οι θεσμοί να λειτουργούν παράλληλα, αλλά να αντιδρούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδρούν και να αναλογίζονται ε, οι μεν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι δε και να τις λαμβάνουν υπόψη. Η, έκθεση αυτή είναι η απάντησή μας στην ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κυριότερος στόχος της έκθεσής μας είναι να τονίσουμε ότι το σημείο αφετηρίας για κάθε θεμελιώδες δικαίωμα πρέπει να είναι ο πολίτης. Πρέπει λοιπόν να ε, είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάθε χρήσιμη πληροφορία στον πολίτη, ούτως ώστε ο πολίτης να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων που του ανοίγονται, των δικαιωμάτων του και των μέτρων που υπάρχουν για την ε, ε, άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Αυτό το σύστημα των θεμελιών δικαιωμάτων πρέπει να είναι χρηστικό για τον πολίτη και τα πάντα εξαρτώνται από την καθημερινή χρήση και χρησιμότητα ε, και αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει έτσι ακόμα πιο αξιόπιστη για τους πολίτες της. Θα πρέπει να ληφθούν ε, μέτρα ε, σε, ε, άμεσα, αλλά επίσης θα πρέπει να υιοθετηθεί μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η κατάσταση των Ρώμα, τα δικαιώματα των παιδιών, η χρήση μειονοτικών γλωσσών είναι ορισμένα μόνο από τα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Και ελπίζω ότι η έκθεση που θα ε, υιοθετήσουμε αύριο θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και στα διάφορα ε, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα και το σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό. Τα θεσμικά όργανα και τα εργαλεία τα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, πρέπει τώρα να ενεργήσουμε. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια, λέει ο Πρόεδρο χαιρετίζω την ε, παρουσία της Επιτρόπου κυρίας Ρέντινγκ, στην οποία δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση σήμερα για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι μόνο διότι λαμβάνει χώρα δέκα χρόνια από την διακήρυξη του χάρτη, είχαμε την επέτειο του χάρτη στην αρχή του μηνός, αλλά επειδή είναι η πρώτη συζήτηση στο Κοινοβούλιο που είναι αφιερωμένη σε αυτό που η συγγήτρια κυρία Γκάλ αναφέρει όσα τη νέα αρχιτεκτονική μετά τη Λισαβόνα. Και έχει δίκιο, αρχίσαμε με μια νέα αρχή, μια νέα εκκίνηση σχετικά με το τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την πολύτιμη συμβολή τους σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε τώρα ένα χάρτη νομικά δεσμευτικό που αποτελεί μέρος πρωτογενούς νομοθεσίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε στην πράξη το χάρτη αυτό και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή υιοθέτησε τον Οκτώβριο την ανακοίνωση για την στρατηγική, για την πρακτική εφαρμογή του χάρτη. Τα ιστόχη κλειδιά της Κομισιόν είναι να γίνουν όσο πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα του χάρτη προς όφελος όσων ζουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών που τους εκπροσωπούν. Ο χάρτης πρέπει να είναι ε, να μας ε, καθοδηγεί η πηξίδα μας, κυρίως όταν νομοθετούμε και αυτό περνάει από την εσωτερική εργασία προπαρασκευής της Επιτροπής ως την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και το Συμβούλιο και μετά στην εφαρμογή των νέων κανόνων από τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή έχει θέσει σε ισχύ μια αξιολόγηση συστηματική της κατάστασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως συνέπεια των νέων νομοθετικών προτάσεων με ε, μια checklist, έναν κατάλογο ελέγχου για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και χαίρομαι που βλέπω ότι η εισήγηση της κυρίας Γκάλ υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση, τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποδώσουν σημασία στην συμμόρφωση προς το χάρτη εκτός της νομοθετικής διαδικασίας, διότι δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα κείμενο επιτάπητος ε, το οποίο ε, έχει συμμορφωθεί προς το χάρτη, όταν ε, τροποποιείται με τροπολογίες αυτό το κείμενο θα πρέπει και ο χάρτης να ληφθεί υπόψη και κάθε όργανο θα πρέπει ε, να βρει πώς θα εξασφαλίσει οι τροπολογίες των νομοθετικών προτάσεων να αξιολογούνται ε, δεόντως. Και γι' αυτό καλό κάνω έκκληση για συνεργασία μεταξύ των οργάνων. Όταν ο νόμος θα έχει γίνει εφαρμοστέως από τα κράτη-μέλη, τότε θα πρέπει να δούμε πόσο ο χάρτης εφαρμόζεται όταν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν νομοθεσία κοινοτική. Και θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι ε, δεν ε, πρόκειται να δηλιάσω ε, να εισαγάγω διαδικασίες επί σε αντίθετη περίπτωση. Έχουμε Επίσης, το θέμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ταχεία προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Σύμβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα για την Κομισιόν και οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται με καλό και επικοδομητικό τρόπο και αν όλα πάνε καλά, όπως φαίνεται, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία στο πρώτο ήμιση του 2011. Λοιπόν, τα πράγματα κινούνται γρήγορα και κινούνται με ικανοποιητικό τρόπο, με αίσιο τρόπο. Επίσης, συμμερίζομαι το στόχο να έχουμε ε, μια αγαστή συνεργασία με τις, ε, τους διεθνείς οργανισμούς. Το κάνουμε αυτό με τον κανονικό τρόπο, με καθημερινό τρόπο. Απλώς ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Η Κομισιό ήδη ε, βασίζεται στην, Ευρωπα... στην ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όταν ε, εκπονεί νέε προτάσεις σχετικά με τα παιδιά. Αυτό έγινε επίσης και για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουμε υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Η εισηγήτρια επίσης μίλησε για τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει ρόλο κλειδί να διαδραματίσει ούτω ώστε να μας δώσει στοιχεία συγκρίσιμα για την κατάσταση στα 27 κράτη-μέλη σε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει. Θέλουμε όχι μόνο ε, να εργαστούμε θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Παραδείγματος χάρη ο οργανισμός θα πρέπει ε, να συμβάλλει στην εργασία της ειδική ομάδας για τους Ρωμά. Ε, θα πρέπει να επεκταθεί η εντολή του οργανισμού τόσο ώστε να μπορεί να παρέχει την πραγματογνωμοσύνη του στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε περιπτώσεις ε, ε, εγκλημάτων και σε αστυνομικές περιπτώσεις. Και γι' αυτό στις 2 Δεκεμβρίου η Κομισιόν υιοθέτησε μια πρόταση τροποποίησης του πολιετούς πλαισίου που αναφέρει τις θεματικές κατηγορίες όπου μπορεί να εργαστεί ο οργανισμός. Και μετά κάτι νέο, κάτι καινούριο που νομίζω ότι είναι τελείωσα σε συμφωνία με τα όσα λέει η συγγήτρια και αυτό είναι η όθηση που δημιουργείται από τη συνθήκη της Λισαβόνας που πρέπει να διατηρήσουμε γι' αυτό την άνοιξη του 2011 η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τον πρώτα ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του χάρτη ε, και αυτό ούτω ώστε κάθε άνοιξη να έχουμε μια τέτοια ετήσια έκθεση η οποία νομίζω ε, θα είναι για το Κοινοβούλιο η κατάλληλη στιγμή ε, για να παρέμβει και να προκαλέσει μια πραγματική συζήτηση για το πώς ο χάρτης υλοποιείται στην πράξη. Και βεβαίως όταν θα ετοιμάσουμε την έκθεση της Άνοιξης 2011, την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή του χάρτη, θα αποδώσω ιδιαίτερη σημασία ε, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά ε, και σε άλλες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα μας επιτρέψει, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο να έχουμε όπως είναι και συνήθεια ε, σε αυτό το κοινοβούλιο, μια συζήτηση για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα μας επιτρέψει να έχουμε κάθε χρόνο μια συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για το ποιο πώς εφαρμόζονται από τα διάφορα κράτη-μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να δούμε πώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκτελούν τα καθήκοντά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ας ακούσουμε τώρα τις ε, παρεμβάσεις εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Σιμών Πουσουτήλ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για τις εκθέσεις της και θέλω να την ευχαριστήσω για το ότι επικεντρώθηκε με τέτοιο τρόπο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Η επικέντρωση ήταν πραγματικά κέρια σημασία για αυτή τη φορά. Θα ήθελα να μιλήσω για τη σπουδαιότητα να εξετάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμελιώδη δικαιώματα για τους πολίτες, για τους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά δεν ερμηνεύουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει να αγνοούμε την έννοια της επικουρικότητας και ότι δεν θα έπρεπε να επικεντρωνόμαστε σε διαφορετικές αξίες των διαφορετικών κρατών μελών. Κάποιοι δυστυχώς όμως χρησιμοποιούν τα θεμελιώδη δικαιώματα για να κάνουν ακριβώς αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να τα αφήσει να αποφασίσουν τα ίδια για θέματα ηθικής, όπως αφορά θέματα ευθανασίας και εκτρώσεων ή αμβλώσεων. Θα έπρεπε επίσης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στα θεμελιώδη δικαιώματα την πραγματική τους σπουδαιότητα, την πραγματική τους σημασία. Δεν θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε δικαιώματα τα οποία δεν είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Κάνω λόγο εδώ και αναφέρομαι σε δικαιώματα όσον αφορά θέματα μετανάστευσης. Πολύ σημαντικά δικαιώματα αυτά, όμως δεν είναι πάντα θεμελιώδη δικαιώματα αυτά. Επίσης θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε συνετές και λογικές θέσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την σημασία της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, για να συμπεράνω, Ολοκληρώνω λέγοντα ότι χρειαζόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμω με ρεαλιστικό πνεύμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουζουτήλ. Παρακαλώ όλου του συναδέλφου να σέβονται τον χρόνο που του έχει δοθεί. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μόνικα Μπενόβα για την ομάδα των Σοριστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, κυρία εισηγήτρια, την κυρία Γκάλ, γιατί πιστεύω ότι ε, εκπλήρωσε τον βασικό στόχο της έκθεσης, δηλαδή ότι καθορίζει σαφώς ε, τους ρόλους των νέων ε, θεσμικών οργάνων και μηχανισμών στα πλαίσια της νέας στρατηγικής μετά τη Λισαβόνα. Τρεις τομείς είναι πολύ σημαντικοί στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Πρώτον, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει όχι μόνο τα δικαιώματα των πολιτών της ή των ατόμων που διαμένουν στην επικράτειά τη. αλλά πρέπει να είναι ο ηγέτη στο θέμα αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πιστεύω στο νέο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νέα υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν να δημιουργήσει μια ειδική υπηρεσία στα πλαίσια της νέας αυτής ε, ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο εξωτερικό. Δεύτερον, πιστεύω ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά τη θέση σε ισχύ της Ειδικής Αφώνας έχουν μια νέα διάσταση πλέον. Γιατί οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νέες δυνατότητες, έχουν τη δυνατότητα πρωτοβουλίας των πολιτών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και τρίτον, πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη για το γεγονός ότι η έκθεση ζητάει από τα κράτη-μέλη να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους, ούτω ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεργασία, το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε και για το ότι η έκθεση αναφέρεται και στην καταπολέμηση της φτώχειας και ε, αυτό είναι κάτι που ζήτησε η πολιτική μας ομάδα. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ρενάτε Βέμπερ για την ε, ομάδα των ε, φιλελεύθερων δημοκρατών. It's on. <laughs> Τώρα λειτουργεί το μικρόφωνο. Συναδελφοί, αύριο το απόγευμα θα μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκόσμια. Σήμερα όμω επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και μετά εκτό από αυτήν. Αυτή είναι η σωστή σειρά πιστεύω εγώ διότι προτού ασκηθούν επικρίσεις σε άλλου, πρέπει να θέσουμε εντάξει τα του οίκου μα Και αν πραγματικά θέλουμε να μα παίρνουν στα σοβαρά δεν πρέπει να αγνοούμε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην επικράτεια της Ένωσης. Αυτό το ψήφισμα για το οποίο θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Κινγκαγκάρ επικεντρώνεται στον τρόπο στο μέλλον για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προαγωγή τους μετά την έναρξη σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Και αυτό δεν αφορά μόνο για το ποιος είναι υπεύθυνο για τι πράγμα, αλλά για τα θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των ανησυχιών μας στο μέλλον. Θέλω μόνο να τονίσω δύο πτυχές εδώ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδα την υποστήριξη στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων για την ιδέα για ένα μηχανισμό παγώματος όπου οι ε, επικρίσεις που ασκούνται σε εθνικές πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν σε πάγωμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτών των διαδικασιών και για μια απόφαση αν θα πρέπει ή όχι να ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο. Ένα τέτοιο μηχανισμό θεωρώ ότι θα δώσει πρόσθετη αξία στο να υπάρχει μια πιο αξιόπιστη πολιτική για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα πλαίσια τη Ένωση. Γι' αυτό ελπίζω ότι αυτό ο μηχανισμό θα μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη όλων των μελών που θα υπερψηφίσουν στην Ολομέλεια όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε αύριο. Η άλλη πτυχή αφορά την υποχρέωση και το δικαίωμα αυτού του Κοινοβουλίου πάντα να, να αναλύουμε τα κράτη-μέλη όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κατονομάζουμε όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις, να κατονομάζονται τα κράτη αυτά. Ευχαριστώ. La parola ora per un e Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Έχει το λόγο τώρα η κυρία Ελέν Φλότρ για την ομάδα των Πράσινων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ καλή εισήγηση, πρώτη μετά τη Λισαβόνα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια την κυρία Γκάλ για την σοβαρότητά της, την, την πνεύμα συνεργασίας, τη διαθεσιμότητά της. Έχουμε τέσσερα μηνύματα. Πρώτον, ε, θέλουμε να ε, εκπληρώσουμε το ρόλο μας με τα νέα μέσα τα οποία διαθέτουμε και με το χάρτη ε, είχαμε τον, την πρώτη πρακτική περίπτωση και η Κομισιόν διένυσε το μισό δρόμο μόνο για την οδηγία της ελεύθερης κυκλοφορίας η Κομισιόν απέφεγε την, ε, την ε, διάκριση δεν θα μπορεί να το κάνει με την επικύρωση από την Ένωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χαίρομαι ε, που θα καλύψει τον υπόλοιπο δρόμο. Η προστιθέμενη αξία αυτής της εισήγησης έγκυται στο γεγονός ότι τονίζει την ανάγκη να ανοιχνεύουμε πρόωρα τα, τις καταστάσεις με ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όταν υπάρχει υποψία τέτοιων παραβιάσουμε και να μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία. Υπάρχει αναγκαιότητα για ένα σύστημα πρόληψης που να εμπνέεται από τον μηχανισμό της περιοδικής καθολικής παγκόσμιας εξέτασης που υπάρχει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει ανάγκη σύνοχης ανάμεσα σε αυτά που γίνονται εντός και εκτός. Η υπογραφή της Συμφωνίας της Κοινοτικής θα είναι πράγματι μια πρόκληση διότι οι πραγματικές διατάξεις αποφασίζονται σε μικτές επιτροπές από τις οποίες αποκλείεται το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία ε, Φλότρ. Ο κύριος Μάνσκι παρακαλώ τώρα από την Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Σας ευχαριστώ πολύ όταν θα αρχίσει να ισχύει αυτή η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα δούμε ότι έχουμε δύο συστήματα προστασίας στην Ευρώπη. Το ένα βασίζεται σε βάση με την ομολογία του ε, ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το άλλο σε σχέση με τις δράσεις και νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Στρασβούργου. Στην έκθεση πρέπει να ε, προβλέπονται οι αντιστοιχίες και η δυνατότητα εκ ερμηνείας και των δύο η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν μπορεί να ερμηνεύεται ότι δημιουργεί μόνο νέε αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, άρθρο, ε, το σχετικό άρθρο το υπενθυμίζει αυτό, αλλά πρέπει να δούμε τα θέματα ποινικού κώδικα και όσον αφορά ε, τα, ε, τους γάμους για παράδειγμα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι εκτρώσεις δεν μπορούν να ρυθμίζονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε δικαστήριο γιατί μια τέτοια πολιτικοποίηση των άρθρων των δικαιωμάτων αυτών μπορεί μόνο να οδηγήσει σε μείωση της εμπιστοσύνης όσον αφορά τα δικαστήρια αυτά. Ευχαριστώ. Και τώρα ε, για την ΚΟΕ, 1,5 λεπτό, η κυρία Μαρή Κριστίν Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της και όλους τους σκιώδεις εισηγητές που συνέβαλαν στην ποιότητα της έκθεσης αυτής, η οποία είναι σημαντική διότι εξάγει τις συνέπειες τις θετικές από την εφαρμογή της Λισαβόνας αν υλοποιηθεί όντως, διότι η υλοποίηση των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιώδης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να αρκεστούμε με τα λόγια. Ε, η συνθήκη, ο χάρτης και η μελλοντική προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορούν να μας προσφέρουν νέα εργαλεία και να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μέλη να διανύσουμε μια νέα περίοδο. Πολλοί λένε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι από τις ουσιαστικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λίγοι έχουν μια ενόραση αδιέρετη και παγκόσμια. Τα δικαιώματα στον χάρτη και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και σε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις ε, που προκύπτουν από την παγκόσμια διακήρυξη έχουν ε, την, το, την ίδια αξία. Δεν υπάρχει πρωταρχία ορισμένων δικαιωμάτων το, το δικαίωμα ύπαρξης έχει την ίδια αξία με την θρησκευτική ελευθερία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ίδια για όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, από την νομική τους κατάσταση. Ξέρουμε ότι το δικαίωμα στην παιδεία, το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, συνέχεια παραβιάζονται και καταπετούνται περίπου σε όλα τα κράτη-μέλη. Η κατάσταση σε σχέση με τους Ρωμά είναι εμβληματική. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να αποφασίσει να προωθήσει διαδικασίες επί παραβάση με τον ίδιο τρόπο όπως για τα οικονομικά αδικήματα. Θα πρέπει να έχουν την ίδια αξία τα δικαιώματα αυτά σε όλο τον κόσμο, στην εξωτερική πολιτική, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει την ίδια σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα οικονομικά διακυβεύματα. Δεν είναι αυτό η περίπτωση. Την Ισία, Λιβύη, Κολομβία, μπορώ να αναφέρω πολλές χώρες. Υπάρχει εδώ ένα θεμελιώδες ε, διακύβευμα ε, και κινδυνεύει η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το μέλλον της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Κριστίνα Μορφάη για 1,5 λεπτό. Ε, magyarként Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως καθώς είμαι Ουγγαρέζα και γυναίκα, πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για το γεγονός ότι μία Ευρωβουλευτήνα Ουγγαρέζα, η κυρία Κίνγκα Γκάλ, ήταν εκείνη η οποία εξεπώνησε αυτή την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά από μια πραγματικά κοπιώδη, εργώδη ε, εργασία. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εργασία αυτή την ευχαριστώ για το ότι υπέβαλε αυτό το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει όμως και ένα γεγονός το οποίο είναι εξόφθαλμο. Πρέπει να τονίσουμε τα πολιτικά και αστικά παραδοσιακά δικαιώματα. Και στην Ουγγαρία είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι εδώ σε σχέση με αυτά τα θέματα στην Ουγγαρία δεν υπάρχει μόνο άσκηση αρνητική διακριτική μεταχείριση ει βάρο μειονοτήτων όπω των συγκάνων. αλλά υπάρχει και η αρνητική αντιμετώπιση του δικαιώματο του συναθρίζεσθε, του εκφράζεστε. Αυτό συνέβη στην Ουγγαρία μεταξύ του 2002 και του 2010. Πρόσφατα η Επιτροπή ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγαρία ενέκρινε συγκεκριμένες ε, αποφάσεις και τοποθετήσεις όπου αναφέρονται τα σχετικά θέματα για να τονιστεί ότι μεταξύ του 2000 και 2010 οι δύο σοσιαλιστικές κυβερνήσεις ποδοπατούσαν διαρκώς και κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω μια ερώτηση προς την εισηγήτρια. Δεδομένη τη σημερινή καταστάσεως ως έχει, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την έκθεση, ακριβώς την έκθεση Τη Επιτροπή ε, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο θα υποβληθεί αυτή η έκθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση και σε σχέση με τα όσα συνέβησαν και έχασαν τη ζωή του στην Ουγγαρία πολλοί άνθρωποι. Θα μπορούσαμε έτσι λοιπόν να υλοποιήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ότι η, η, η, η Πολιτικών Δικαιωμάτων ήταν ακριβώ. Ε, ένα άτομο το οποίο είχε συμμετάσχει σε αυτές τις δράσεις στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους άλλους ε, γεγραμμένους ομιλητές, ξεκινώντας από τον κύριο Σαλβατόρη Γιακολίνο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε με ικανοποίηση μια έκθεση ε, σαν αυτή που με τόση σύνεση συνέταξε η συνάδελφος Γκάλ η οποία καταγράφει με πολύ συγκεκριμένο και λεπτομερή τρόπο την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για το θέμα αυτό και την εφαρμογή του θα ήθελα συντομία να εκφράσω ορισμένες σκέψεις. Για τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που τώρα είναι υποχρεωτικός, είναι νομικός ε, δεσμευτικός με τη ε, συνθήκη της Λισαβόνας, θα έπρεπε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι η προστασία ε, των ατόμων περνάει από περνάει σε μια συγκεκριμένη ε, πολιτική με την οποία συμφωνούν όλοι και θα έχουμε έτσι συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις διατάξεις της Λισαβόνας και της Οχόλμης και να σκεφτούμε τα θέματα της ε, αλληλεγγύης και ε, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και βεβαίως η αρχή της επικουρικότητας δεν μπορεί να είναι περιορισμός για την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τους πολίτες. Έχουμε το νέο ε, κανονισμό που αφορά την ε, πρωτοβουλία ε, των πολιτών και αυτό, όλα αυτά αποτελούν το νέο πλαίσιο, ε, το νομοθετικό. Όλα αυτά έχουν συγκεκριμένο στόχο να ε, δοθεί ε, αξία στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όσον αφορά τους ελέγχους και τις αποτελεσματικές κυρώσεις, αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2013 που είναι το έτος ε, της ηθαγένειας, ευρωπαϊκό έτος ηθαγένειας. Με αυτή την ε, ευκαιρία θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα αποτελέσματα να επιδείξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάικλ Κάσμαν έχει το λόγο. Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Στην Ευρώπη μπορεί κανείς να, έχει διακριτική μεταχείριση ότι είναι γυναίκα. Όταν ε, ε, ε λόγω της ηλικία του, του σεξουαλικού προσανατολισμού για την ε, ε παροχή υπηρεσιών ε, ε, αν είναι κανείς ε, παντρεμένος με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή με απλή συμβίωση μπορεί να τύχει διακριτικη μεταχείρισης με βάση την επικουρικότητα επίσης. Έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. σε, κάποιοι συμμετέχουν και κάποιοι όχι. Βλέπουμε, καθόμαστε εδώ και βλέπουμε να, να έρχεται η ξενοφοβία, ο, η ομοφιλοφοβία και κοιτάξτε τι έγινε και με τους Ρωμά. Δεν διδαχτήκαμε τίποτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή από τη δεκαετία του 30 όταν κλείσαμε τα μάτια μας και δεν κάναμε τίποτα για αυτούς που ήταν διαφορετικοί από εμά. Δεν βλέπουμε ότι η θρησκεία χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να αυξηθεί ε, η διακριτική μεταχείριση. Ε, και σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να δούμε ότι το να περιορίζονται τα δικαιώματα ενός άλλου σημαίνει ότι περιορίζονται τα δικά μας δικαιώματα. Ε, δεν έχουμε τίποτα για να, που να μας κάνει περήφανους. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Ντάνιελ Βαντενστούπ. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ρίχνει νέο φως στα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα προσχωρώντας ε, στην σύμβαση ε, θα υπάρχουν ε, δικαιοδοσίες οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές. Πώς θα γίνει η αξιολόγηση αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρήσει στη σύμβαση μπορεί να βρεθούμε σε ναρκοπέδιο. Ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω μια ερώτηση στην Επίτροπο. Ε, ένα ένταλμα ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται για την υπόθεση Κονταϊβέλ ε, σε 290 σε 23 το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής είναι ανώτερο από το γενικό συμφέρον. Η απόφαση αυτή με εκπλήσει. Θα ήθελα να μου πει τι πιστεύει η Επίτροπος για αυτήν την δικαστική απόφαση και ποιος είναι ο αντίκτυπος του χάρτη πάνω στην μελλοντική νομοθεσία. Ευχαριστώ κύριε Βαντεστούπ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μίλαν Σβέρ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για μια εξαιρετική έκθεση. Αληθεύει πράγματι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια νέα πλέον κατάσταση που σημειώνεται και διαμορφώνεται στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επεκτείνουμε το πεδίο της ελευθερίας και αυτό είναι εξαιρετικό. Κάνουμε λόγο για μια τρίτη γενναία δικαιωμάτων. Όμως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνει εξίσου και την επανόρθωση αδικιών του παρελθόντος. Στην έκθεση κάνουμε λόγο για τη νέα γενεά δικαιωμάτων. Αγνοούμε και ξεχνάμε όμως ε, θέματα όπως αποκατάσταση και ε, επιστροφή ε, της κυριότητας και ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων που είχαν κατασχεθεί από ένα προηγούμενο καθεστώς ή τα θύματα στη δεκαετία του 1940 σε αρκετές κέντρο-ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε εμείς μια που προσαρμόζει πολιτικές αποφάσεις σε αυτή τη συγκυρία. Και είναι δική μας ευθύνη να επανορθώσουμε τα σφάλματα και τις αδικίες του παρελθόντος. Μόνο όταν θα έχουμε κάνει αυτό το πράγμα θα έχουμε καθαρή τη συνείδηση για να μιλάμε για μια τρίτη γενεά δικαιωμάτων για το παρόν και το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κίνγκα Γκόντς για ένα λεπτό τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τη συνθήκη της Λισαβόνα ε, μεταμορφώθηκε και πήρε υποχρεωτικό δεσμευτικό χαρακτήρα. Μπορούν να ξεκινήσουν κοινοτικέ διαδικασίε σε περιπτώσει παραβιάσεων και παραβάσεων. Υπάρχουν και κοινωνικέ επιπτώσει σαν συνέπεια τη κρίση στα κράτη-μέλη και αυτό οδηγεί σε περιορισμό των δικαιωμάτων αντί σε επέκτασή του, Περιορίζονται τα μέσα του τύπου, τα δικαιώματα στην απεργία, στο κοινωνικό διάλογο, τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων. Αυξάνεται η κοινωνική διακριτική μεταχείριση περιορίζονται τα δικαιώματα συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θεματοφύλακα των Συνθήκων έχει την υποχρέωση να αντιδράσει σε δεδομένων αυτών των σημάτων. Έχουμε εδώ και πρόταση για να υπάρξει η δράση επιτρόπου αρμοδίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και θα πρέπει εδώ να τοποθετήσετε όταν ε, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να μην υπάρχει μόνο το θέμα ανάλυση ε, από πλευρά των υποψήφιων κρατών μελών αυτών των δικαιωμάτων, αλλά και των Ευχαριστώ, κυρία Γκόνς. Η κυρία Μόνικα Λουίζα Μακοβέη έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Κίνγκα για την έκθεσή της. Έχουμε τώρα μια κοινότητα αξιών και αρχών που αντικατοπτρίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό περιλαμβάνει και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι η πιο σύγχρονη κωδικοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, τηρούν τον χάρτη αυτό όταν εφαρμόζουν την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διατάξει του χάρτη είναι άμεσα εφαρμοστέ από τα εθνικά ε, δικαστικά συστήματα που έχουν τώρα μεγαλύτερε εξουσίε. Δεύτερον, έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και την ε, δικονομία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και ε, ε, επίση την διασφάλιση των δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης μπορούμε να έχουμε προστασία των δικαιωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε επίπεδο εθνικού εθνικού δικαίου. Επίσης πρέπει να παρακολουθούμε τις αποφάσεις του ε, Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εφαρμόζουν άμεσα μέσω των δικών του θεσμικών οργάνων τι διατάξεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν ε, νομικούς και ε, θεσμικούς μηχανισμούς. Το βασικό ζήτημα όμω είναι η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων για τα θύματα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ε, η κυρία Ιωάννα Ζενίσιν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι. Η συμπερίληψη της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης ε, ε, δεν είναι εκείνο το οποίο εξαντλεί τις αρμοδιότητες της ε, Ένωσης ε, διότι αποτελεί πραγματικά μέρος των αρμοδιοτήτων μας αυτό και γι' αυτό καλώ τις πολωνικές αρχές να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να τηρήσουν αυτή τη χαρτά. Δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα ή καμία άλλη δικαιολογία. Είναι μόνο μια πολιτική απόφαση που έχουν λάβει που βλάπτει τους πολίτες. Η υιοθέτηση της χάρτας είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά και την επόμενη μελλοντική ε, προεδρία. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα άσχετα ποια είναι η χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους. Δυστυχώς στην Πολωνία δεν το κατανοούν αυτό ακόμα και όσον αφορά και τα δικαστήρια. Ένα ειδικό πρόβλημα είναι εδώ η αρνητική διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών βλέπουμε ότι πρέπει με κάθε τρόπο να εφαρμοστούν τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της βίας ε, κατά των γυναικών. Εδώ πρέπει να αρχίσει η δράση μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άνταμ Κώσα για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαν αρκετές παρεμβάσεις που τόνισαν τις πιο διαφορετικές ε, σημαντικές ε, πτυχές της έκθεσης. Έχουμε ενώπιόν μας εν τέλει μια έκθεση που συμπεριλαμβάνει όλα τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς να τονίζει κάποια ξεχωριστά ε, δικαιώματα εις βάρος των άλλων. Και για μένα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και με ικανοποιεί ιδιαίτερα, διότι τονίζεται η μάχη κατά των ανισοτήτων και προάγεται η ισότητα. Η προαγωγή αυτής της έκθεσης, ε, ο στόχος της είναι η προαγωγή των θεμελιδών δικαιωμάτων. Το κύριο τμήμα της παρέμβασής μου αφορά αυτό ακριβώς το τμήμα, δηλαδή το σεβασμό και την υλοποίηση της χάρτας. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να το καταφέρουμε. Αυτό θα γίνει αν αναγνωρίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Και επίσης ότι θα πρέπει να υποφελούνται από ίση μεταχείριση όλοι οι πολίτες. Αν κάποιος, οποιοδήποτε, για κάτι το οποίο δεν είναι δική του ενοχή ε, γι' αυτό διώκεται και υφίσταται αρνητική μεταχείριση πρέπει να τύχει της ανάλογης βοήθειας και συνδρομής για να μπορεί να υποφεληθεί πλήρως από τα δικαιώματα του πολίτη ακριβώς όντας ένας πολίτης ίσως με τους άλλους. Είναι μια μακρά διαδικασία, είναι μια εργόδης προσπάθεια, απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια σίγουρα και η διαδρομή είναι μεγάλη. Η έκθεση της κυρίας ε, Κίνγκα Γκάλ είναι ένα ορόσημο, ο μύτος της Αριάδνης ε, προς αυτή την πορεία και γι' αυτό χαίρομαι και εκφράζω την ικανοποίησή μου γι' αυτό. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τη διαδικασία Catch the Eye και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ε, λάβει 11 ε, ονόματα συναδέλφων που θέλουν να μιλήσουν. Για λόγους χρονικού περιορισμού δεν μπορούμε να δεχτούμε και τους 11. Μόνο 6 αιτήματα τέτοια μπορούμε να δεχτούμε. Προφανώς με τη σειρά που έχουν υποβληθεί και ε, λαμβάνοντα υπόψη την έκφραση όλων των πολιτικών ομάδων, ε, ζητώ λοιπόν συγγνώμη από του συναδέλφου που δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Η κυρία Άννα Ζαρμπόσκα για ένα λεπτό είναι η πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να επισημάνω έναν κίνδυνο κυρίως ε, ο συνδυασμός των διαφόρων μορφών καταπολέμησης των διακρίσεων μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις. Αυτό αναφέρθηκε ήδη ε, στην Βιέννη την περασμένη εβδομάδα στην συνάντηση του ESC. Αν αυτό ε, γίνει νομίζω θα υπάρξουν διακρίσεις κατά των ατόμων. Βλέπουμε πως αυτή η έννοια των διακρίσεων μεταβάλλεται, αλλάζει πρόσωπο. Αν υπάρχει μία προσπάθεια πάνω στην οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούμε, θα πρέπει να είναι να επανέλθουμε ε, στην αρχική έννοια της λέξης διάκριση. Νομίζω ότι ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να παίξει κρίσιμο ρόλο από την άποψη αυτή και πρέπει να ελέγχουμε επίσης την λειτουργία αυτού του οργανισμού. Ή αλλιώς ε, θα είναι απλώς ε, ένα, μια επιβάρυνση οικονομική όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για ολόκληρη την Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία εισηγήτρια έκανε εξαιρετική δουλειά. Ωστόσο από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ουγγρική παροιμία που λέει ότι αν κάτι δεν γίνεται, ε, είναι, δεν, δεν είναι χρήσιμο, είναι περιττό σαν τα πέταλα ενός ε, ψόφιου αλόγου. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασίες προσφυγής ε, σε περίπτωση παραβιάσεων και παραβάσεων. Έχετε μεγαλύτερο θάρρος κυρία Ρέντινγκ από όλους τους άνδρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το θάρρος να υψώσετε το ανάστημά σας ενώπιον του κυρίου Σαρκοζή, πράγμα που δεν έκανε ο κύριος Μπαρόζο εδώ και πολύ καιρό. Μεγάλη μεγάλες προκλήσεις είναι αυτές που αντιμετωπίζονται τώρα, διότι η Ουγγρική κυβέρνηση που θα αναλάβει την μελλοντική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιόρισε τα πολιτικά δικαιώματα, κατάργησε τα δικαιώματα των συνδικαλιστών και των κρατικών υπαλλήλων και δεν σέβεται και την προστασία της, ιδιωτικής προστασ... Ε, της προσωπικής ιδιοκτησίας. Όταν αφαιρεί από 3 εκατομμύρια άτομα Ούγγρους πολίτες ε, τις ε, αποταμιεύσεις τους, τα όσα είχαν στις Έχετε το θάρρος κυρία Ρέντινγκ. Ξεκινήστε αυτή την προσφυγή βάρο βάρος της Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σόνια Αλφάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα άρθρα 6 και 7 ε, της συνθήκης, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία παραβιάζεται η ελευθερία του τύπου, τα κόμματα συμμετέχουν σε εκλογές με ψεύτικες υπογραφέ, υπάρχει εμπλοκή με τη μαφία ε, ε, ε, και τον Πρωθυπουργό που ελπίζουμε ότι δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα. Όλα αυτά που ακούμε μέσω του Wikileaks. Γι' αυτό το λόγο ε, θα ήθελα ε, να ε, ζητήσω υποστήριξη της τροπολογίας που αφορά τις παραγράφους 20 και 40 και που αφορά τις παραβιάσεις σε εθνικό επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξάλλου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την παραβίωση των θεμελιδών δικαιωμάτων και τέλος η υπάρχει ε, το πρόβλημα των ε, μειονοτήτων, της ελευθερίας τύπου ε, και για όλα αυτά που σας λέω ζητώ να καταψηφιστεί η έκθεση. Η κυρία Φιγκερέντο τώρα έχει τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Διατηρείται όπως γνωρίζουμε Πολλέ φορές ε, με πολλούς τρόπους η αρνητική διακριτική μεταχείριση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αυτό πλήττει αρκετές κατηγορίες ε, πολιτών και πολιτισμικές ε, μειονότητε. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε μια αρνητική μεταχείριση γενική που υφίσταται ει βάρος των γυναικών. Η αρνητική μεταχείριση των γυναικών διατηρείται στις πιο διαφορετικές, στα πιο διαφορετικά επίπεδα με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα έλεγα και μάλιστα σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι γυναίκες εργαζόμενες εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες να έχουν πρόσβαση στην εργασία. Εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες να προβιβαστούν στη σταδιοδρομία τους και εξακολουθούν να είναι θύματα της μισθολογικής ανισότητας και που πάντα πλήττουν τις γυναίκες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν υπολογισμοί που λένε ότι 18% είναι η μισθολογική εις βάρος των γυναικών αρνητική μεταχείριση το μειονέκτημά τους μισθολογικά. Πρέπει κάτι να γίνει να καταπολεμηθούν αυτές οι ανισότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρανς Ομπερμάγια έχει το λόγο. Πρόεδρε, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, δίνει τον κίνδυνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποφασίζουν για οτιδήποτε αμφιβάλλω αν είναι πάντα α, αμερόληπτες αυτές οι αποφάσεις. Ε, όταν έχουμε εδώ περιπτώσεις ε, τον άσυλο ε, μεταναστών και τα Και βλέπουμε εδώ ότι κάποιοι συντάκτες ετοιμάτων προσπαθούν στο δικαστήριο αυτό να οδηγήσουν στο πάγωμα της συμφωνίας, του Δουβλίνου και να εκδοθούν ή να καταλήξουν στην Ελλάδα. Γιατί, διότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης που ε, κλειδονίζει τα θεμέλια της Ευρώπης. Αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τέτοιου είδους ε, έλλειψη σεβασμού ε, έχει για τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε τέτοιες αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Μεσάρος. Κύριος Μεσάρος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν ικανή να ασκεί επικρίσεις εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά έλλειψη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην δική μας περίπτωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Τώρα όμως άλλαξε η κατάσταση. Έχουμε και τα στοιχεία αυτά τα οποία εκτίθενται στην έκθεση Kinga Gal. Χρειάζεται ένα σύστημα προστασίας των θεμελιωδών θεμελιδών δικαιωμάτων που μπορούμε να αναπτύξουμε σήμερα χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεν μπορούν να παραμένουν ατιμόρυτα τα θέματα παραβιάσεων και παραβάσεων των δικαιωμάτων των πολιτών μα. Πρέπει να καταλήγουν σε δικαστικέ προσφυγέ και σε διεκδίκηση των δικαιωμάτων για επανόρθωση δικαστικά. Πρέπει να ασκείται προσφυγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλε τι δικαιολογημένε περιπτώσει. Επιπλέον, όταν επιβαρύνονται με προσκόμματα και δυσκολίε τέτοιου είδου προσφυγέ, πρέπει τόσο περισσότερο αυτή η δυνατότητα προσφυγής να ασκείται για να προστατεύονται πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα. Πρέπει να τερματιστεί η αρνητική ε, διακριτική μεταχείριση και να προστατεύονται και τα μειονοτικά δικαιώματα στις μειονοτικές γλώσσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η τελευταία ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα, θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο επίπεδο των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν και να επιλύονται. Τα κράτη-μέλη πρέπει εδώ να επομίζονται την ευθύνη. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να εκπονείται μια στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα δικαιώματα των παιδιών είναι σημαντικά διότι αυτό λείπει στο διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής ε, εκμετάλλευσης των παιδιών και της κακοποίησής τους. Ένα άλλο θέμα είναι τα θέματα τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, ε, διότι πολλές φορές είναι και αυτά θύματα αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Είναι σημαντικό να εκπονούνται και να υπάρχουν στρατηγικές για την προστασία των ατόμων με μειονεξία και ειδικέ ανάγκες. Επίση, η κατάσταση των παιδιών και των γυναικών και αυτή είναι ευάλωτη. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινωνικά συνοδευτικά μέτρα για να προστατεύονται τα άτομα αυτά κατά του κοινωνικού, από τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις ανισότητες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλα τα μέλη της Επιτροπής που εργάστηκαν για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλους τους ευβουλευτές που έλαβαν μέρος ε, σήμερα σε αυτή τη συζήτηση εδώ δείχνοντας ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα κατέχουν σημαντική θέση. Και δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω τα όσα λέχθηκαν από πάρα πολλούς ευρωβουλευτές ότι δηλαδή ήρθε η κατάλληλη στιγμή να ασχοληθούμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια αξιοπιστία. Επίσης και να μπορούμε να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε παραμιλήσει λίγο το θέμα αυτό. Δεν θα είναι η κατάσταση ίδια στο μέλλον. Το γεγονός ότι θα έχουμε μια φορά το χρόνο βάσει της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του χάρτη πράγμα που περιλαμβάνει περίπου όλες τις παρατηρήσεις και τα θέματα που αναφέρθηκαν από τους μεν και τους δε σχετικά με ειδικέ διακρίσεις. Αυτό θα είναι για μας η στιγμή όπου πράγματι θα μπορέσουμε να θέσουμε επιτάπητος όλα τα θέματα, να δούμε τι δεν λειτουργεί καλά και να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. πώς ε, να διορθώσουμε τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η ιδέα του freezing mechanism, όπως το υπενθύμησε η συγγήτρια, αυτό το σύστημα πρόληψης ε, όπου θα μπορούμε να παρέμβουμε σε μια δράση συγκεκριμένη σε ένα κράτος μέλος ε, όταν αυτή η δράση δρομολογείται. Είπα στους εμπειρογνώμονες μου να αναλύσουν ένα τέτοιο μηχανισμό και τα θέματα τα θεσμικά σχετικά με ένα τέτοιο μηχανισμό είναι πάρα πολύ περίπλοκα για την ώρα, αλλά θα πρέπει ακόμη να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο τα πράγματα, αλλά για την ώρα μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να μπορέσουμε να δράσουμε με τον τρόπο αυτό και ότι θα χρειαζόταν μια τροποποίηση συνθήκης για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό πρόληψης. Η ιδέα είναι ελκυστική. Θα συνεχίσουμε να έχουμε διαβουλεύσεις για να δούμε ποιος μηχανισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς αλλαγή μεταχείρισης για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα επίγοντα θέματα. Θα ήθελα ωστόσο να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε κάτι ε, σε ένα σφάλμα που γίνεται συχνά, ότι δηλαδή ο χάρτης δεν μπορεί να εφαρμοστεί με απόλυτο τρόπο. Εφαρμόζεται, ισχύει μόνον όταν τα κράτη-μέλη ε, ε, θέτουν στην πράξη ευρωπαϊκούς κανόνες. Όταν δηλαδή μια οδηγία ευρωπαϊκή που έχει αποφασιστεί ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, μετά εντάσσεται, ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Τότε ο χάρτης ισχύει, αλλά δεν ισχύει έτσι εν κενό. Ε, δηλαδή σε όλες τις άλλες ε, περιπτώσεις τα εθνικά δικαστήρια έχουν την ευθύνη παρεμβάσεως. Τη στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα υπάρξει μια άλλη διάσταση, μια συμπληρωματική διάσταση πρόσθετη ε, που θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε στην πράξη με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την πολιτική των δικαιωμάτων. Αυτό που μου φαίνεται πρωταρχικής σημασίας πέραν από όλα τα ειδικά θέματα τα οποία τέθηκαν και στα οποία θα απαντήσω ε, μεμονωμένα και προσωπικά στους βουλευτές που τα έθεσαν, νομίζω ότι το μεγάλο θέμα, η μεγάλη υπόθεση είναι η θεμελιώδης υπόθεση. Προς τα έξω, στα κράτη-μέλη μας, στις κυβερνήσεις, δεν, ξέρω, δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί πραγματικά ε, τη σημασία του χάρτη. Έχουμε συνεπώς μια μεγάλη εργασία ενημερωτική να εκτελέσουμε, ούτως ώστε παντού να υπάρξει αυτή η κουλτούρα των δικαιωμάτων, αυτή η πολιτική των αξιών, ούτως ώστε παντού όλοι να διαρωτόμαστε όταν ε, θεσπίζουμε ένα νόμο, όταν εφαρμόζουμε ένα νόμο, αν αυτός ο νόμος είναι σύμφωνος με τις αξίες τις οποίες έχουμε προσυπογράψει. Αυτός ο, ο αυτοματισμός θα έλεγα περίπου, όταν ως ηθήνοντες πολιτικοί δρούμε, θα πρέπει πάντοτε να διαρωτόμαστε αν αυτά τα οποία πράττουμε είναι σύμφωνα, είναι σύμβατα με τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, τα οποία έχουμε υιοθετήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ε, τέλειο στοιχείο, αν θέλετε. Και μπορώ να σας πω ότι σήμερα η Επιτροπή θα λάβει μια απόφαση σχετικά με την κατάργηση της εξεκουατούρ, δηλαδή θα υπάρξει μια πρόταση ούτω ώστε οι αποφάσεις της δικαιοσύνης να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα παντού στην Ευρώπη. Οι ε, σημαντικές αποφάσεις και για πρώτη φορά ε, κατά τη διάρκεια της πρότασης αυτής ε, της νέας ρύθμισης έχουμε ελέγξει αν αυτή η απόφαση θα είναι σύμφωνη με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο μια ανάλυση οικονομική, όχι μόνο ένα impact assessment, μια ε, αξιολόγηση του αντικτύπου στην αγορά, αλλά ένα impact assessment για το τι επίδραση θα έχει αυτή η απόφαση σχετικά με τις αξίες. Βλέπετε ότι σιγά σιγά οδεύουμε προς αυτή τη νέα πολιτική και νομίζω ότι θα έπρεπε ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να προσπαθήσουμε ούτω ώστε αυτή η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του χάρτη να γίνει μια μεγάλη στιγμή αλήθειας όπου θα θέσουμε επιτάπητος εγώ ως Επιτροπή με την έκθεση που θα παρουσιάζω και εσείς ως Κοινοβούλιο με τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσετε, θα αποκριθείτε, θα κατακρίνετε ή θα χαιρετήσετε αυτήν την έκθεση θα είναι η μεγάλη στιγμή όπου πραγματικά θα χαιρετησετε αυτη την εκθεση θα ειναι η μεγαλη στιγμη οπου πραγματικα θα δειξουμε στον εξωτερικό κόσμο, στους ψηφοφόρους μας ότι ναι, ο χάρτης είναι ζωντανός. Δεν είναι μόνο ένα κείμενο, θα είναι μια πρακτική και αν δεν γίνει μια πρακτική ή αιρετή ε, του λαού θα το πούνε δυνατά. Αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε, να δημιουργήσουμε κατά τη διάρκεια των δύο ή τριών ετών πριν από τις επόμενες εκλογές. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σιγά σιγά με την άνοιξη, με την πρώτη έκθεση, με την πρώτη άσκηση αυτού του είδους και μετά θα υπάρξει μία παράδοση που ε, θα εγκατασταθεί εδώ, σε αυτόν τον οίκο, ούτω ώστε κανείς να μην μπορεί να πει όταν την Τετάρτη και την Πέμπτη θα ασχοληθείτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός των συνόρων της Ένωσης ότι δεν έχετε βάλει σε τάξη το δικό σας το σπίτι. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα η συγχύτρια κυρία Κίνκα Γκάλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για τα λόγια που υποστήριξαν και ενθάρρυναν εμένα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Επίτροπο για αυτό το ανοιχτό πνεύμα και συνεργασία που μας έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστούμε επικοδομητικά και για τα συγκεκριμένα θετικά μηνύματα που μας έδωσε. Πιστεύω ότι υπό το πρίσμα των σκιωδών εισηγητών όλα όσα επιθυμούσαν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση και γι' αυτό η διαδικασία ήταν αποδεκτή. Δεν μπορώ λοιπόν να υποστηρίξω και να δεχτώ τις τροπολογίες που τώρα έχουν εκ νέου κατατεθεί στην Ολομέλεια διότι πιστεύω ότι όσα έχει τώρα η έκθεσή μου είναι πλέον αποδεκτή από όλους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μέσα στο Γενικό Σύστημα Προστασίας των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν έρχεται η ώρα να προστατευτούν αυτά δεν είναι δυνατόν να χάνουμε την ουσία προσπαθώντας να δούμε κάποιες Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στα συγκεκριμένα θέματα, να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις και να πάρουν χειροπιαστά μορφή και να γίνουν χειροπιαστά δικαιώματα και πραγματικότητα. Γι' αυτό ελπίζω ότι αύριο στην Ολομέλεια θα υλοποιηθούν όλα αυτά και θα υιοθετηθούν και η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα και το θέμα των παιδιών, θα ληφθούν υπόψη, καθώς επίσης και η αποδοχή της πρωτοβουλίας των πολιτών. Ένα αποτέλεσμα που δίνει την δυνατότητα να κάνουμε πραγματικά λόγο για μια Ευρώπη των πολιτών, με μια ε, τέτοια πτυχή δημοψηφίσματος ή πολιτικής πρωτοβουλίας από πλευρά των πολιτών. Ελπίζω ότι αύριο λοιπόν έτσι θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα περάσουμε μετά και στην εξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικαιωμάτων παγκόσμια. Θα πρέπει να εξεταστεί από την ε, Ουγγρική Προεδρία αυτό το θέμα στο μέλλον. Θέλω να τονίσω όμως κυρίες και κύριοι ότι εμείς εδώ σε αυτό το σώμα πρέπει να αποφύγουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Και αυτό θέλω να το πω σε εκείνου και στρέφομαι στους ε, ε, Ούγγρους σοσιαλιστές σε εκείνου που ήταν μάρτυρες παραβιάσεων και μάλιστα των πιο σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τώρα όμως δίνουν μαθήματα, υψώνουν το δάκτυλο και κάνουν κατήχηση και μαθήματα. Ιδιαίτερα όταν έχουν οδηγήσει εκείνοι στο να έχουν χάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσοι πολίτες. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στι 12.30. Περνάμε τώρα στην εντολή Ευρωπαϊκή στην Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, ε, έκθεση Τερέζα Χιμένες. Παρακαλώ, κύριε Γκάσμαν, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ε,